Και έτσι ολοκληρώσαμε την συνεδρίαση. Τα πρακτικά θα τα λάβετε για έγκριση στην επόμενη, για την επόμενη σύνοδο. Και τα ψηφίματα τα οποία εγκρίθηκαν θα α, διαβιβαστούν στους υπεύθυνους. Κύριε Οντή, θέλετε το λόγο. Oui, Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Παρεμβαίνω επί τη βάση του εσωτερικού κανονισμού, αλλά ξεχνάω αυτή τη στιγμή το άρθρο. Προβλέπει το τον Ευρωπαϊκό Ύμνο όταν υποδεχτούμε κάποιον ε, σε επίσημη επίσκεψη. Πρόσφατα μας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Τινησίας, ο, πρόεδρο, ε, ε, πρόεδρος του Ισραήλ, Σιμών Περές, και δεν ακούστηκε ο, Ευρωπαϊκός Ύμνος. Τι γίνεται, για ποιο λόγο και να εκφράσω και τη λύπη μου που δεν ακούστηκε ο Ευρωπαϊκός Ύμνος αυτές τις δύο ευκαιρίες στο ημικύκλιο. Κύριε Οντή, δεν θυμάστε το άθρο του κανονισμού και εγώ δεν θυμάμαι αν το έχουμε αλλάξει αυτό. Θα το κοιτάξουμε. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Θα συμπεριληφθεί αυτό στα πρακτικά. Διακόπτεται η σύνοδος και σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό και καλή επιστροφή.